Αναλόγως. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Χαουτάλα προστασία έναντι των επιδοτούμενων εισαγωγών από χώρε που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε στη δεύτερη έκθεση Χαουτάλα, προστασία έναντι εισαγωγών από μη ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βαλένσα. Συμφωνία σύμπραξη στο τομέα της βιώσιμης αλίας μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας της Λιβερίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση ΜΑΤΟ. Συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξης ΕΕ Μαυριτανίας. Αλλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπουονάνο. Συμφωνία συνεργασία για το μη στρατιωτικό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγηση με την Κορέα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τόμασιτς νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχή 2014-2020. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Sven Giegold. Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Μπλοκ υπαριθμών 1. Διαδικαστικό, κύριε Κάρβερ, έχετε. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρατήρησα ότι έχουμε 25 σελίδες ε, τροπολογιών που κατέθεσε ο εισηγητής χθες το βράδυ, στα γερμανικά κιόλας. Ε, γίνεται ε, λόγω της πληροφορία του Ηνωμένου Βασιλείου ή να ξέρουμε κάτι για τη γλώσσα που θα επικρατήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Πρόεδρος, εμένα μου είπαν ότι οι τροπολογίες υποβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και έχουν μεταφραστεί όλες και δεν καταλαβαίνω το νόημα των σχολείων σας εκτός από το, ε, το σχόλιο που θέλετε να ακουστεί για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα μήνα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την έκθεση Κίκουλ. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Ηλιάνα Γιώτοβα για την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 16 κατά τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22 αρχικό κείμενο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 46 αρχικό κείμενο κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 53 αρχικού κειμένου ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 56 αρχικό κείμενο δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. Παράγραφος 63, αρχικό τμήμα, αρχικό κείμενο, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 68, αρχικό τμήμα, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη. Ερχόμαστε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Θα περιμένουμε λίγο να φύγουν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως και γρήγορα. Καλή σας όρεξη.